Ε, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε τις εργασίες μας. Έχω ένα άσχημο νέο. η δολοφονία του Jean Serge Νερά, Γάλλου αστυνομικού από την ΕΤΑ. Το πρόβλημα της τρομοκρατίας δεν έχει λυθεί. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια εκ μέρους όλου του Κοινοβουλίου στην οικογένεια του αστυνομικού. Ελπίζω να βρεθούν και οι δολοφόνοι αλλά και οι εντολή της δολοφονίας. Επίσης, άλλο άσχημο νέο, στην Κούβα συνελήφθησαν 30 διαδήλωτες ε, της ομάδας ε, Woman in White. Πρόκειται για μητέρες ε, και συζύγους μελών της αντιπολίτευσης που κρατούνται. Αυτές οι γυναίκες έχουν βραβευθεί με το βραβείο Ζαχάροφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς τις υποστηρίζουμε αυτές τις γενναίες γυναίκες Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, κοινή συζήτηση για δύο εκθέσεις. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την κατάσταση του ευρώ. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Τσικλούνα και την έκθεση Sven Giegold για την ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ευρώ και των δημοσιονομικών το 2009. Το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Έντουαρτ Σικλούνα. Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια ήταν, αποτελούσαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως θεματοφύλακα της ε, νομισματικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Στην ετήσια